Well, good evening. Let us start the meeting. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλωσορίζω τα μέλη και το ακροατήριο στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Φορολογικά μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή δεν αδρανούσε, μια αντιπροσωπεία μας πήγε σε αποστολή στη Ουάσιγκτον τον Ιούλιο. Και άλλη αντιπροσωπεία πιο πρόσφατα πήγε στην Λετωνία. Και έτσι πήραμε πρώτο χέρι πληροφορίες και στοιχεία για πολλά από τα στοιχεία που μας αφορούν. Θα συζητήσουμε ψηφιακή φορολόγηση σήμερα. Όλοι ξέρουμε ότι η αδελφή μας Επιτροπή, η ΕΚΟΝ, ασχολείται με δύο νομοθετήματα. Στόχος τους η εξασφάλιση ότι οι ψηφιακές εταιρείες δεν ξεφεύγουν όσον αφορά τη φορολόγηση. Στην αποστολή μας στην Washington, D.C., η ψηφιακή φορολόγηση ήταν από τα θέματα που ενδιέφερε τους ομολόγους μας. Ήταν πολύ ζωηρές συζητήσεις. Η ακρόαση θα ωφεληθεί από τη γνώση που αποκόμισαν να τις συζητήσει στα μέλη μας. Με τη σημερινή συζήτηση θα εφαρμόσουμε την εντολή μας συμβάλλοντας τις συζητήσεις περί φορολογήσεως της ψηφιακής οικονομίας. Είμαι πεπισμένος ότι η σημερινή συζήτηση θα τροφοδοτήσει το έργο των νομοθετικότητες οίκων στο σχετικό τομέα. Η ακρόαση θα αποτελεστεί από δύο παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων. Ο ένας είναι από τον ΟΣΑ και δύο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Έντουαρτ Φολσόντας από την Γενική Διεύθυνση Ταξούντ θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνοδεύεται από τον κύριο Βάτ Βαν Ράιν από την DG ε, Taxud. Ο κ. Έρικ Ρομπέ από τον ΩΣΑ θα παρουσιάσει τη θέση του φορέα για την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Καλώς ήρθατε κύριοι στην συνεδρίαση. Θέλουμε να ακούσουμε τις παρουσιάσεις σας. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας σχετικά με την ψηφιακή φορολόγηση. Κάθε θεσμικό όργανο θα έχει ένα δεκάλεπτο για παρουσίαση. Μετά την παρουσίαση από τους ομιλητές θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής υπό τη μορφή ερωταπαντήσεων. Κύριε Φολσόγκας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Μπάρτ και εγώ είμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προετοιμάζουμε το πακέτο για την ψηφιακή φορολόγηση. Δοθέντων των χρονικών περιορισμών, θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε κάποια σημεία, τις βασικές πτυχές του πακέτου. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που συζητούνται. Αν κάποια από τα θέματα δεν καλυφθεί στην παρουσίασή μου, παρακαλώ να με ειδοποιήσετε και να το τονίσετε σε ερωτήσει. Θα καλύψω ακροθυγώς το πρόβλημα προς επίλυση. Μετά ακροθυγώς θα περιγράψουμε τις λύσεις που διαφαίνονται και που προτείνουμε. Να τονίσω κάτι. Είναι το ίδιο πρόβλημα. Επιλύεται από διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι θέλουμε να λύσουμε. Τη φορολόγηση εισοδήματο εταιριών και πώς εφαρμόζεται η φορολόγηση στο ψηφιακό τομέα. Έχουμε ψηφιοποίηση, που είναι ένα γεγονός, και επιτρέπει σε όσοι βαθμίδες της κοινωνίας να κινητοποιηθούν ψηφιακά. Αυτό είναι πολύ καλό. Ενθαρρύνουμε την ψηφιοποίηση. Και η ψηφιακή ενία αγορά είναι πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σαν πολίτες, σαν χρήστες, Όλοι δεχόμαστε ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει ωφέλη. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και τις εταιρείες και τους κανόνες για φορολόγηση των εταιριών που έχουν θεσπιστεί πριν από 100 χρόνια και περισσότερα για, τις, για τη φορολόγηση επιχειρήσεων και αυτοί οι κανόνες εδράζονται επί της ενίας της φυσικής παρουσίας. Δηλαδή μια εταιρεία πληρώνει άμεσα φόρους στη δικαιοδοσία, σε μια δικαιοδοσία αν είναι φυσικά παρούσα εταιρεία εκεί αν έχει έδρα εκεί, μόνιμη παρουσία εκεί, διότι πριν από 100 χρόνια βλέπετε, αν μια εταιρεία ήθελε να κινηθεί σε μια αγορά, έπρεπε να είναι φυσικά παρούσα, να έχει μια αποθήκη, να ανοίξει ένα κατάστημα. Γι' αυτό οι κανόνες βασίζονται πολύ επί της φυσικής παρουσίας. Αν συνδυάσουμε τις δύο πραγματικότητες, τι βλέπουμε, ότι δεν ταιριάζουν. Τα ψηφιακά επιχειρησιακά μοντέλα έχουν διάφορα χαρακτηριστικά σε αόρατα, σε άειλα υλικά, παράγουν την αξία, άειλη αξία. Και κλίμακα χωρίς μάζα, όπως λέει ο ΩΣΑ. Δηλαδή, από μακριά μπορεί να παρέχει υπηρεσίε και να πλησιάζει τον καταναλωτή από μακριά. Οι ψηφιακέ επιχειρήσει δεν έχουν έδρα για φορολόγηση σε μια δικαιοδοσία, συγκεκριμένη δικαιοδοσία, ενώ κινούνται επιχειρηματικά σε αυτή τη δικαιοδοσία και ωφελούνται από τις υποδομές ε, της ε, δικαιοδοσίας χωρίς να φορολογούνται από αυτή τη δικαιοδοσία. Γι' αυτό λέμε ότι το πλαίσιο τη φορολόγηση εταιριών είναι κάτι απερχιωμένο και οι ψηφιακέ επιχειρήσει δεν μπορούν να πληρώσουν φόρο εισοδήματο εκεί που ε, επιχειρούν, λόγω των κανόνων που βασίζονται φυσική παρουσία. Όλε οι λύσει που προτείνουμε στο πακέτο ψηφιακή φορολόγηση προσπαθούν να επιλύσουν το ίδιο πρόβλημα από διαφορετική γωνία και σε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Εδώ βλέπετε ότι τα προβλήματα που αναφέρουμε αναπτύσσονται, αυξάνονται. Γνωρίζετε το πολιτικό πλαίσιο, δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα αυτά. Συζητούνται εκτενώς. Εξετάστηκαν από τον ΩΣΑ είχαμε πολιτική εντολή από το Συμβούλιο να τα επεξεργαστούμε και εμείς και να υποβάλουμε προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου το Μάρτιο. Προτείνουμε λοιπόν αυτές τις λύσεις. Το πρόβλημα που περιέγραψα είναι παγκοσμίου εμβελίας και γι' αυτό χρειάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο η λύση. Τι εννοώ με αυτό. Μια λύση που θα συμφωνηθεί σε επίπεδο ΟΣΑ, σε διεθνέ επίπεδο. Ε, ξέρουμε ότι αυτή η σφαιρική λύση χρειάζεται χρόνο για να είναι λογική. Είναι περιπλοκότατο το ζήτημα, βλέπετε. Η δομική λύση που πιστεύουμε που είναι η μόνη συνεπάγεται επαναπροσδιορισμό βασικών ενιών ε, μόνιμη εγκατάσταση κλπ. που φορά τη φορολόγηση των εταιριών. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν τους κανόνες για την φορολόγηση των εταιριών σε επίπεδο της Ένωσης και προτείνουμε οδηγία για να αλλάξουν οι κανόνες που ισχύουν μεταξύ κρατών μελών και έχουμε και συστάσεις να αλλάξουν οι κανόνες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών πρέπει να καθορίσουμε εκ νέου τους κανόνες για τη φορολόγηση εταιριών λαμβάνοντας υπόψη τον ψηφιακό παράγοντα. Δύσκολο το εγχείρημα. Χρειάζεται χρόνο. Γι' αυτό προτείνουμε βραχυπρόθεσμη λύση. Ε, προσωρινή λύση. Να εφαρμοστεί μέχρι την πλήρη λύση που θα εφαρμοστεί. Προσωρινό μέτρο. Ο, η φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Η πλήρης λύση, θα την αναφέρω οδηγό αυτήν, έχει στόχο να αλλάξει την απάντηση σε δύο ερωτήσει. Αυτό που μας κάνει να έχουμε δύο ερωτήσει. Όταν θέλουμε να καθορίσουμε τι φόρο πληρώνει μια, μια εταιρεία σε ένα κάτω Τι φορολογούμε και πού το φορολογούμε. Για να πληρώσει άμεσους φόρους, εταιρικούς φόρους μια εταιρεία σε μια χώρα πρέπει να έχει φορολογική σχέση με αυτή την νομοθεσία. Αν βασίζεται η εταιρεία στη φυσική παρουσία, ε, δεν υπά... αν δεν είναι φυσική παρουσία δεν υπάρχει αυτός ο φορολογικός δεσμός. Γι' αυτό προτείνω να δημιουργηθεί μια σχέση ψηφιακής φορολόγησης η εταιρεία για να, να πρέπει να καταβάλει φόρους σε ένα κάτω μέλος δεν είναι κάτι, δεν είναι απαραίτητο να έχει ψηφιακή, μόνο να έχει ψηφιακή μόνιμη παρουσία, αλλά θα πρέπει και τα κέρδη να μπορούν να σχετιστούν με αυτή τη μόνιμη ε, παρουσία, την ψηφιακή της εταιρείας σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό προτείνουμε να λάβουμε υπόψη την ψηφιακή πτυχή των επιχειρήσεων με τον τρόπο, στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει την κατανομή των κερδών. Αυτά βλέπετε. Τι προτείναμε. Πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια. Και από τη στιγμή που θα έχουμε καθορίσει ότι υπάρχει η ψηφιακή φυσική παρουσία, θα πρέπει να γίνει κατανομή των κερδών σύμφωνα με τη λειτουργική ανάλυση που χρησιμοποιείται τώρα, ενεργητικό κίνδυνος που αναλαμβάνει η εταιρεία και ψηφιακή πτυχή, κάτι που λείπει σήμερα. Πάω τώρα στο προσωρινό μέτρο. Αυτό που περιέγραψα, η πλήρης λύση, η τελική λύση, που πιστεύουμε ότι θα δώσει τα ακριβέστερα αποτελέσματα και θα είναι η ακριβέστερη λύση του προβλήματος, θα είναι μια ε, συμφωνία, θα χρειάζεται μια δύσκολη συμφωνία πρώτα. Εν τω μεταξύ έχουμε πιέσεις που ασκούνται πάνω μας να δράσουμε για προσωρινά μέτρα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης της φορολογικής βάσης στα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάποια αδικία που διαπιστώνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες όσον αφορά τους κανόνες περιφορολογήσεως διότι εντάσσονται στα παραδοσιακά κριτήρια αυτές οι εταιρείε και διαμαρτύρονται. Συναντήσαμε αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείε και μας είπαν ότι είναι σε μια θέση δύσκολη, δυσχερή, μειονεκτική επιχειρηματική, διότι αντιμετωπίζουν άλλε εταιρείε που δεν έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν παίζουν με του ίδιου κανόνε. Έχουμε κατακαιρματισμό τη ενιαία αγορά, οπότε έχουμε και πρόβλημα συμμόρφωση. Αρκετά έχουν αρχίσει να θεσπίζουν προσωρινά μέτρα και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί ότι οι προσωρινέ λύσει αποτελούν πραγματικότητα και χωρί δράση Ευρωπαϊκή Ενώση, ποιο είναι ο κίνδυνο. Ότι θα καταλήξουμε σε εμβαλωματικέ λύσει 28 προσωρινών μέτρων. Γι' αυτό προτείνουμε έμεσο φόρο, δυνάμει του άρθρου 113, όσον αφορά τα μεικτά κέρδη μέσω που προέρχονται μέσω ε, κάποιων ψηφιακών δραστηριοτήτων και μόνο. Μετά, γιατί προτείνουμε κάτι τέτοιο θα τεθεί και το θέμα του, της φορολόγησης κύκλου εργασιών. Αυτός απορρέει από τη φορολόγηση των κερδών και των εισοδημάτων των εταιριών. Γιατί προτείνουμε ένα φόρο κύκλου εργασιών. Αν θέλουμε προσωρινό μέτρο το οποίο εφαρμόζεται τώρα, η αντιμετώπιση των κενών και διαφορών όσον αφορά τους κανόνες φορολογής εταιριών, αυτό το μέτρο το προσωρινό δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τους κανόνες που θέλουμε να αλλάξουμε και η φορολόγηση εισοδήματο θα έχει τους ίδιου περιορισμού που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Μέσω μιας τελικής λύση. Τέλος. Αυτό το προσωρινό μέτρο έχει, είναι πολύ στοχευμένο και από πλευρά των φορολογητών φορολογουμένων ατόμων, φυσικών προσώπων που πρέπει να καταβάλουν το φόρο και από πλευρά δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το νέο φόρο. Φορολογούμε μόνο κάποιες ψηφιακές δραστηριότητες που βασίζονται πολύ στη συμμετοχή του χρήστη. Αυτή η συμμετοχή του χρήστη έχει νομισματική αξία, χρηματική αξία και είναι τη βασική εισρωή για την παραγωγή κέρδους εισοδήματος από Θέλουμε αυτό το δυναμικό να το αναγνωρίσουμε και γι' αυτό ο φόρος εφαρμόζεται σε αυτές τις δραστηριότητες με υψηλή ε, συμμετοχή των χρηστών και όχι σε άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστώ κύριε Φορσόγκας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μας παρουσιάσετε ποια είναι η προσέγγιση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω τώρα το λόγο επίσης στον άλλο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας κάνει και αυτό στην παρουσίαση του. Με συγχωρείτε, θα ακολουθήσει ο κύριο Ρομπέρα από τον Όσα. So, um, as introduction, given... Um... Θα ξεκινήσουμε μία εισαγωγή. Θα σας παρουσιάσω λίγο τα όσα έχουμε κάνει στα πλαίσια του πλαισίου για τα BEPS στον Όσα, δηλαδή για τις προκλήσεις που δημιουργεί τη φορολόγηση ή η ψηφιοποίηση και ο ψηφιακός κόσμος. Ξεκινήσαμε με το πρώτο ε, BEPS, γνωρίζοντας πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί είχαμε μια σειρά από φορολογικά σκάνδαλα που μας οδήγησαν στην προσπάθεια δημιουργίας φορολογικού ε, πλαισίου για τις πολύ ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις. Το 2014 λοιπόν η πρώτη προσπάθεια με πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε το 2015 και η προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε πως δεν έχει κλείσει, πως χρειάζεται να δούμε και κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη φοροαποφυγή και έχουμε ε, μία νέα ομάδα οργασίας η οποία ονομάζεται Task Force για την ψηφιακή οικονομία με νέα εντολή το 2016 και 2017 στα πλαίσια του ε, πλαισίου για τα BEPS ε που είναι το νέο βήμα στο οποίο παρακολουθούμε και εποπτεύουμε το πώς ε, τα σχετικά μέτρα εφαρμόζονται. Και πρέπει να σας πω πως εδώ έχουμε πια σήμερα πάνω από 117 μέλη, τα οποία εργάζονται σε ισότιμη βάση. Στα πλαίσια αυτής της νέας εντολής, η Task Force συνέχισε τις προσπάθειές της με μία προθεσμία η οποία αρχικά είχε μπει για το 2020, μετακινήθηκε και είπαμε ότι θα βρούμε κάποιες λύσεις για τα δυσεπίλητα πρόβλημα, τα οποία ήδη ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε σε μία ενδιάμεση έκθεση τον Μάρτιο του 2018. Και θα σας παρουσιάσω εντάχει κάποια από τα συμπεράσματα. Πριν όμως μπούμε σε αυτά, θα ήταν χρήσιμο να μπούμε στην πρώτη έκθεση του 2015 για τα BEPS, στα συμπεράσματα εκεί και στα ευρήματα τα οποία δημιούργησαν το έδαφος στο οποίο τώρα εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε το πλαίσιο. Το πρώτο έβριμα είναι πως δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κλάδος οικονομίας που να είναι η ψηφιακή οικονομία. Είναι μια διαδικασία μεταμόρφωσης ολόκληρη της οικονομίας, οπότε δεν μπορούμε να περιχαρακώσουμε ε, κάποιες επιχειρήσεις και κλάδους λέγοντας πως φορολογικά αυτά θεωρούνται ψηφιακή οικονομία. Δεύτερον, όταν εξετάζουμε τα διάφορα πλαίσια που δημιούργησαν όλες οι υψηλά ψηφιοποιημένες εταιρείε, διαπιστώσαμε πως οι τεχνικές που χρησιμοποιούν λογιστικά κτλ. είναι αρκετά διαφορετικές ε, από αυτές που έχουν οι άλλες μία ψηφιοποιημένε εταιρείε. Παρ' όλα αυτά έχουν και πάρα πολλά κοινά στοιχεία και αυτό αποτελεί την κοινή βάση κρίσης για τα BEPS και είπαμε ότι στην πρώτη ε, έκθεση για την ε, ε, ψηφιακή οικονομία με το πρόγραμμα πλαίσιο όπου μιλάμε για την ψηφιακή μεταμόρφωση και την ψηφιοποίηση, τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Δηλαδή, τότε καταλήξαμε στην παραδοχή πως η ψηφιοποίηση και τα σχετικά ε, χαρακτηριστικά τα οποία παρουσίασε προηγούμενος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή η μεγάλη εξάρτηση από τα άϊλα, η χρήση ε, και η εκμετάλλευση των δεδομένων των χρηστών για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, όλα λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ δεν δημιουργούν θέματα BEPS, ουσιαστικά οξύνουν κάποια από τα προβλήματα αυτών, ε, κυρίως ε, λόγω φορολογικών τακτικών που ακολουθούνται έτσι ώστε να αποφεύγουν τη φορολόγηση. Είπαμε λοιπόν πως υπάρχουν κάποια, ε, κάποιες προκλήσεις φορολογικές που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής και των μέτρων, αλλά ε, θέματα που εμπίπτουν στην ίδια τη φύση αυτών των επιχειρηματικών μοντέλων, δεν είναι τόσο ηθικά ζητήματα, αλλά κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα για τα οποία αναρωτιόμαστε αν το τρέχον φορολογικό πλαίσιο για άμεση και ήμιση φορολογία θεωρείται ακόμα ικανό. Και είπαμε πως αυτές οι βασικές προκλήσεις θα πρέπει να απαριθμηθούν, να περιγραφούν ε, και για την άμεση αλλά και για την έμεση φορολόγηση. Για την έμεση όπως ξέρετε και εσείς έχουν ήδη προκριθεί κάποιες λύσεις και είχαν σχεδιαστεί από τότε και σήμερα έχουμε πια για το ΦΠΑ, για παράδειγμα, κάποιε παγκόσμιε λύσει, οι οποίε εφαρμόζονται σε γενικέ γραμμέ από πολλά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., λόγω των σχετικών με τον ΦΠΑ ε, αλλά και άλλε 60 χώρε που σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμόζουν τι παγκόσμιε αυτέ ε, λύσει για το θέμα του φόρου προστιθέμενη αξία. Ξέρω πω τα γνωρίζετε. Εδώ το πρόβλημα είναι η αποτελεσματική συλλογή στη χώρα κατανάλωσης όταν ο πάροχος υπηρεσίας ή ψηφιακού προϊόντος δεν βρίσκεται, ε, δεν έχει φυσική παρουσία στην χώρα κατανάλωσης. Για την άμεση φορολόγηση και το κομμάτι εκεί, αντιμετωπίσαμε το εξή πρόβλημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί. Και νομίζω ότι αυτά εξήγησε και προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησε για κατανομή κερδών, για τον έξους, για τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται σε σχήματα τα οποία εντάσσονται στο τρέχον φορολογικό πλαίσιο. Δηλαδή, ποιος έχει το δικαίωμα φορολόγησης και ποιος κατανέει με τα δικαιώματα αυτά. Αυτό δεν ήταν έντολη της Task Force, αλλά ε, θέλαμε να δούμε το θέμα αυτό, της κατανομής δικαιωμάτων φορολόγησης και συμφωνήσαμε πως χρειάζεται παραπάνω δουλειά στους κλάδους αυτούς, έτσι ώστε ε, αργότερα να δοθεί και εκεί μια λύση. Εδώ δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα, αλλά η συμφωνία ήταν να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Uh, Έχουμε και μια νέα εντολή για το πακέτο. Και εδώ τα κομβικά σημεία σχετίζονται με τις ευρύτερες ε, προκλήσεις στην άμεση φορολόγηση που επαναλαμβάνω κατά τη διάρκεια του Project PEPS δεν βρήκαν μια λύση. Και για να έχουμε μια συνενετική προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε, το πιο σημαντικό ήταν καταρχήν να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα για το τι συμβαίνει και μετά να παρακολουθήσουμε όποιες σχετικές εξελίσεις έχουμε και που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, όπως επίσης και με τον τρόπο από τον οποίο οι επιχειρήσει χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα των εργασιών που φέραμε σε πέρας και που βρίσκονται στην ενδιάμεση έκθεση, δηλαδή εδώ γίνεται μια ανάλυση των επιχειρηματικών μοντέλων, γιατί είναι μοντέλα τα οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ψηφιοποιημένα και επίσης παρακολουθήσαμε την εφαρμογή των BEPS και τις επιπτώσεις που έχει σε εισρωές, εκροές στα επιχειρηματικά μοντέλα και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα ε, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το κομμάτι της φόρου αποφυγής και βέβαια να παρακολουθήσουμε τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη με την ψηφιοποίηση, με τις προκλήσεις σε φορολογικό επίπεδο. Ξέρετε πως αρκετά κράτη έχουν υποβάλει προτάσεις σαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό το, η πρόκληση της ψηφιοποίησης. Και αρκετά κράτη, όπως η Ινδία για παράδειγμα, έχει την, ε, ε την εξισωτική εισφορά ε, που ισχύει. Και ο στόχος είναι να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση εμείς για το ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις και να δώσουμε τη δυνατότητα κάποιου πρόοδου έτσι ώστε να επιτευχθεί συνένεση για μια μακροπρόθεσμη λύση. Ε, σημαντικό σημείο σε αυτή την ενδιάμεση έκθεση από φέτος το Μάρτιο ήταν η δημόσια διαβούλευση που οργανώθηκε στην Καλιφόρνια. Με μεγάλη συμμετοχή από ενδιαφερόμενους από πολύ διαφορετικές ε, προελεύσεις. Και βέβαια όλη η διαδικασία αυτή και η νέα εντολή και τα παλαιότερα BEPS έχουν ε, γίνει υπό την αιγίδα του ε, πλαισίου SDG 20 που εγκρίνει τις διάφορες φάσεις των ευρημάτων και ανανεώνει τις εντολές της Task για την ψηφιακή οικονομία. Η πιο πρόσφατη έγκριση είναι αυτή τη ενδιάμεση έκθεση του Μαρτίου του 2018 η, η Προεδρία Αργεντινής. Περνάμε τώρα στην ενδιάμεση έκθεση. Εδώ έχουμε 8 κεφάλαια που καλύπτουν πάρα πολλά διαφορετικά θέματα και πιστεύω πως ίσως εδώ το πιο σημαντικό είναι να τονίσουμε το τι έχουμε κάνει ήδη για τις ευρύτερες φορολογικές προκλήσεις και βλέπετε εδώ τα διάφορα θέματα που έχουμε εντάξει στην ενδιάμεση έκθεση και αν κοιτάξετε δεξιά, που είναι θέματα φορολογικής πολιτικής, θα διαπιστώσετε πως καταρχήν σημειώθηκε πρόοδος στη διερεύνηση των προκλήσεων αυτών και των συνεπειών των βασικών χαρακτηριστικών της α, ψηφιοποίησης για το φόρο εισοδήματος. Έχουμε την εξάρτηση από τα άειλα, την συμμετοχή χρηστών, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν προεκτάσει που επηρεάζουν τα φορολογικά και τα κράτη έχουν δει το θέμα αναγνωρίζοντας πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι διαφορετικές οι απόψεις για το τι θα πρέπει να γίνει με την ψηφιοποίηση και με τα διάφορα στοιχεία πληροφορικής που χρειάζεται κάθε διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο για να, για να λειτουργήσει. Οι θέσει των κρατών, όπως βλέπετε εδώ, για τις ψηφιακές επιπτώσεις για τη φορολογία εισοδήματος, είναι αυτές που εμπίπτουν στις διάφορες κατηγορίες και έχουμε τρεις κατηγορίες κρατών που εμείς εντοπίσαμε. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτές οι χώρες που θεωρούν πως το πρόβλημα σχετίζεται με ένα από τα χαρακτηριστικά της ψηφιοποίησης που είναι η χρήση, η συμμετοχή των χρηστών. Και εδώ χρειάζεται στοχευμένες αλλαγές ε, στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο, αλλά το αφήνουν εκεί μια δεύτερη ομάδα κρατών που θεωρεί πως η ψηφιοποίηση είναι ένα σύμπτωμα απλώς ενός μεγαλύτερου προβλήματος που το προκαλεί η παγκοσμιοποίηση και κάποιες από τις βασικές αρχές της τρέχουσας φορολογικής πολιτικής δεν είναι ε, αρκετά εξελιγμένη για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Άρα λοιπόν οι προκλήσεις δεν περιορίζονται στις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να δοθούν αποκρίσεις σε ευρύτερα προβλήματα, οπότε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί γενικότερα σε όλη την οικονομία. Και τρίτη κατηγορία κρατών που θεωρεί ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που να σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και όταν εφαρμοστούν τα BEPS θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Εδώ είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει δέσμευση από όλα τα κράτη στο πλαίσιο ανεξάρτητα με το σε ποια ομάδα κρατών που περιέγραψαν ανήκουν και έχουν δεσμευθεί να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να βρουν μια μακρόπρόθεσμη λύση που θα ε, αλλάξει και τους κανόνες κατανομής ε, κερδών αλλά και τα όσα σχετίζονται με τον έξους. Και θα κλείσω λέγοντας πως νομίζω πως μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το κατά πόσο είναι βιώσιμη η πρόοδος το κλάδο αυτό γιατί θεωρούμε πως έχουμε την τελική προθεσμία του 2020 και μία από τις βασικές χώρες που, θα είμαι ειλικρινής, ε, προσπαθούσε να μπλοκάρει ε, την πρόοδο στις συζητήσεις αυτές, γιατί ε, διαφωνεί με την διάγνωση που κάνουμε και για τον τρόπο που βλέπουμε την ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση, ή είπα, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει στο να συζητηθούν τα θέματα αυτά και έχει δεσμευθεί μαζί με τις υπόλοιπε χώρες, ζητώντας να γίνει μια τροποποίηση στη, στους τρέχοντες κατε, κανόνες κατανομής κερδών και νέξους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Και εδώ, στην τελευταία διαφάνεια, εντοπίζουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα σε επίπεδο task force. Και ποιο είναι το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα εργασίας, για να πετύχουμε συνένεση για μακροπρόθεσμη λύση, Κάποιε τεχνικέ λοιπόν εργασίε για το τι, θα πρέπει, τι μορφή θα πρέπει να έχει αυτή η μακροπρόθεσμη λύση. Σα ευχαριστώ πολύ. Open the for questions. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρομπέρ για την παρουσίαση της θέσης του ΩΣΑ. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Θα Γίνουν τώρα οι ερωτήσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν διάρκεια πέραν του ενός λεπτού. Και θα δώσω καταρχήν το λόγο στον εισηγητή του ΕΛΚ, τον κύριο Νίντερμαγερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μας για την παρουσίαση αυτή. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την ακρόση που είχαμε στην ΕΚΟΝ Πιστεύω ότι εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μία πιο δίκαιη κατανομή της φορολόγησης. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ουσιαστικά μπορεί να δημιουργηθεί διπλή φορολόγηση. Είτε αν θέλετε την φορολόγηση ενός υπάρχοντος ε, κέρδους το οποίο έχει ήδη φορολογηθεί, υπάρχει αυτή, αυτός ο κίνδυνος και βάσει ποιων στοιχείων θα γίνεται η εκτίμηση. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι εδώ δεν πρόκειται μόνο για την ψηφιακή οικονομία, αλλά και παραδείγματος χάρη ε, τις πωλήσει ε, εξ και άλλου είδους εμπορικές συναλλαγές και όχι μόνο την ψηφιακή οικονομία. Συμφωνείτε? Και όσον αφορά την κατανομή του κέρδους είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η σωστή κατανομή του κόστους. Είναι ίσως λίγο πιο γενική η ερώτησή μου. Πώς μπορούμε να καθορίσουμε το κόστος και τη βάση κόστους για αυτήν την νέα ε, ίδρυση, αν θέλετε, φορολογικής βάσης. Ευχαριστώ. Κύριε Ρομπέρ, θέλετε να απαντήσετε. Μπορώ να σχολιάσω το δεύτερο σημείο της παρέμβασής σας. Νομίζω ότι όσον αφορά τη διάβρωση της ε, φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών. Υπάρχουν ε, πολλές χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και που θεωρούν ότι ουσιαστικά η ψηφιακή οικονομία αυτό που κάνει είναι ότι υπερβάλλει και μεγιστοποιεί υπάρχοντα προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό, μια σημαντική ομάδα ε, χωρών που κάνει αυτή τη διαπίστωση. Αν συμφωνείτε, αν και εσείς κάνετε αυτή τη διάγνωση, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν λύσεις βραχυπρόθεμες και πιο μακροπρόθεσμες. Καταρχήν, εντοπισμός των συγκεκριμένων ε, χαρακτηριστικών μιας αγοράς, χαρακτηριστικά που αφορούν μια χώρα ή μια αγορά, συγκεκριμένοι τρόποι για να υπάρξει τροποποίηση του υπάρχοντος πλαισίου και μέτρα για να φτάσουμε σε μια πιο δική κατανομή ε, της ε, φορολογίας και τέλος να εντοπιστούν οι αδυναμίες του συστήματος, του σημερινού συστήματος, έτσι ώστε να υπάρξει πιο δίκαιη φορολόγηση στο μέλλον και να πάψουν να υπάρχουν τα κενά και οι αδυναμίες που σήμερα επιτρέπουν αυτές ε, τις ε, στρεβλώσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε πρόσβαση σε μια αγορά, να μπούμε σε μια αγορά και ενδεχομένως να συζητήσουμε τις διάφορες ε, εναλλακτικές λύσεις και λύσεις βραχυπρόθεσμες ή πιο μακροπρόθεσμες. Ευχαριστώ πολύ, Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα που κάνατε. Εγώ συμφωνώ. Δεν θέλουμε να φορολογήσουμε περισσότερο, αλλά διαφορετικά και αυτό ουσιαστικά με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο, δηλαδή να αλλάξουμε τους υπάρχοντες κανόνες έτσι ώστε να ενσωματωθεί η νέα ψηφιακή οικονομία και τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και με τα μεσοπρόθεσμα, τα προσωρινά αυτά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί. Θέλουμε να κανονίσουμε με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο, καταρχήν το γενικότερο πλαίσιο, τις αγορές που ε, σήμερα λειτουργούν, τις εταιρείες που έχουν φυσική παρουσία, δεν έχουν φυσική παρουσία, δημιουργούν κέρδος και να βασίσουμε την φορολογία και στη φυσική παρουσία αλλά και στην ε, φορολόγηση των κερδών. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι γιατί θα πρέπει εδώ να ισχύουν οι κανόνες αυτοί και στις ε, εσωτερικές αγορές, στις εθνικές αγορές. Όπως ξέρετε, η συνθήκη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αυτό, de facto, οδηγεί όμως σε διακρίσεις. Γι' αυτό και θα πρέπει εδώ να χρησιμοποιήσουμε και τις ε, εθνικές αγορές, τις εσωτερικές αγορές, έτσι ώστε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για να πάψουν να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις, να επιτρέψουμε δηλαδή στις ε, ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις αλλά και σε παγκόσμιους ομίλους να συνυπολογίσουν όλες τις δραστηριότητες τους εντός και εκτός των συγκεκριμένων αγορών που φορολογούνται. Το θέμα τώρα της ύπαρξης των αξιόπιστων στοιχείων, βεβαίως εδώ όλες οι χώρες δεν επιτρέπουν την επιβολή αυτών των κανόνων και το θέμα της επιβολής ενός ευρωπαϊκού φόρου, μιας ευρωπαϊκής φορολογίας σε μια μη ευρωπαϊκή επιχείρηση, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Μια αμερικανική εταιρεία, ινδική, κινέζικη εταιρεία. Θα πρέπει ουσιαστικά να είναι κατανοητό στον Ευρωπαίο καταναλωτή ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να καταβάλουν των ΦΠΑ στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να υπάρχει μια απλοποιημένη διαδικασία τύπου one-stop shop, μια διαδικασία διαφανής και απλή, έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές να μην δυσκολεύουν την ε, ίσπραξη του φόρου, την κατανόηση των κανόνων και σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά τα οποία πάνω από 750 εκατομμύρια συγκεκριμένα. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θέστε κάποιες ερωτήσεις. Συνεισηγητής για το S&D. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Από το τελευταίο ερώτημα, για να είμαι ακριβής, Πολύ συχνά ακούγεται το εξή επιχείρημα. Ότι έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι υπάρχει παράκαμψη της φορολογήσεω από τις ψηφιακέ εταιρείε που είναι εκτό της Ευρωπαϊκής Ενώση, εδρεύουν εκτός αλλά δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση με το Facebook να συνεχίσει να, να πουλά τι υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την θέσπιση αυτών των διατάξεων χωρίς να υπόκειται στην ψηφιακή φορολόγηση. Νομίζω το απαντήσατε, αλλά είναι μια ερώτηση που τίθεται συχνά. Άλλο ένα επιχείρημα που συχνά ακούγεται κατά της ψηφιακής φορολογήσεως. Τι γίνεται με τις μη ψηφιακές εταιρείες. Δηλαδή αρχή της φορολόγησης στον χώρο που παρέχεται υπηρεσία στον πελάτη μπορεί να γίνεται χωρίς να υπάρχει μια ψηφιακή παρουσία. Μπορείτε να μας πείτε αν η προτασή τη φορολόγηση ψηφιακή υπηρεσία θα ισχύει και για παραδοσιακέ εταιρείε μη ψηφιακέ, όπω οι φαρμακευτικές εταιρείε ή αυτέ που παράγουν άλλα φυσικά προϊόντα, παιχνίδια, φεριπίν ή ενδύματα. Και τέλος προς τον ΩΣΑ, τον κύριο Ρομπέρ. Ήσασταν πολύ αισιόδοξο όσον αφορά την κοινή δράση και τη συμφωνία και συνένεση μεταξύ χωρών του ΟΣΑ μέχρι το 2020. Πού βασίζεται η, φιλο... αισιοδοξία σας. Ε, ελπίζω να έχετε δίκιο. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να προστατεύσει την κυριότητα τη ενία αγοράς, να εξασφαλίζει θεμητού όρου, ισότιμού όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφευθεί η διάβρωση της φορολογητέας βάσεως μέσω των προτάσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως το συζητάτε αυτό και στα πλαίσια του, των συζητήσεων του ΟΣΑ, της προσωρινής διατάξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω την τελευταία ερώτηση. Πού θα εφαρμοστεί αυτή η φορολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών. Θεμελιώδες θέμα. Δεν είναι φόρος επί εταιριών συγκεκριμένων ή επί ομίλου εταιριών, δεν είναι φόρος που αφορά συγκεκριμένο τομέα, ούτε φόρος επί ψηφιακών εταιριών. Όπως είπατε σωστά, μπορεί να έχετε και παραδοσιακή εταιρεία που παρέχει κάποιες υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο του DST. Είναι ένας φόρος ο DST που πρέπει να καταβάλλεται από φορολογούμενα πρόσωπα βάσει κριτηρίων και που παρέχουν κάποιες ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες καθορίζονται καλά στην οδηγία. Διαφημιστικές υπηρεσίες, μια μετάφραση πώληση στοιχείων. Αν πάρουμε μια φαρμακευτική εταιρεία, Φερρυπίν, παραδοσιακή εταιρεία, που πολλή στοιχεία, όχι οποιαδήποτε στοιχεία, στοιχεία που καθορίζονται σαφώς από την ομοθεσία που παράγονται από τους χρήστες μέσω ψηφιακών πλατφορμών κλπ. Αυτή η εταιρεία εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογή του DST. Για την πρώτη ερώτηση, δεν την έπιασα καλά. Δεν κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ της δικής σας ερωτήσεως και του προηγούμενου Ευρωβουλευτού. Πώς θα παρακάμπτουν οι εταιρείε ενδεχομένως τη φορολόγηση. Ο κίνδυνος είναι ελάχιστος και δεν είναι χειρότερος από τη δυνατότητα που η ίδια έχει δυνατότητα να παρακάψει τον φόρο που ήδη έχει καθοριστεί τώρα, που ισχύει τώρα. Οι φορολογικές δικαιοδοσίες πρέπει να έχουν ένα μηχανισμό για να καλύπτουν αυτούς τους κινδύνους και να ελαχιστοποιούν τους εν λόγω κινδύνους και θα το ενδεχόμενο. Ευχαριστώ, Όσα. Uh, a few words on the um, Θέλω να πω δύο λόγια για το θέμα του κατά πόσο είμαστε αισιόδοξοι για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στα πλαίσια του All-Inclusive Framework και κυρίως στο ότι διαπιστώνουμε να υπάρχει ε, μία νέα δυναμική. Έχω ξεκινήσει με το project αυτό το 2013 και το παρακολουθώ έκτοτε, δηλαδή έχουν πέρασει πάνω από πέντε χρόνια και πρέπει να σου πω πως η δυναμική άλλαξε στην Task Force, οι ισορροπίες άλλαξαν και δεν ξέρω βέβαια ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, δεδομένης στις νέες ε, θέσης που έχουν λάβει κάποια κράτη. Για τις ε, μονομερείς δράσεις και κυρίως για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ψηφιακό φόρο υπηρεσίας, αν δείτε τα δικά μας μέλη δεν υπάρχει συνένεση για το κατά πόσο χρειάζεται μια άμεση και μονομερής δράση στο σημείο αυτά. Και δεν μοιάζει να είναι πιεστική αυτή η ανάγκη. Και τώρα, εκ μέρους του ΟΣΑ, να σας πω πως θεωρούμε πως το δικό μας DNA βρίσκεται το να πετυχαίνουμε πολυμερείς συνενετικές λύσεις. Οπότε έχουμε μία φυσική αποστροφή προς τις μονομερείς και μη συντονισμένες μεταξύ τους δράσεις. Πολλές από τις χώρες που ανήκουν στη Task Force, εκτός από αυτές που είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουν με συμπάθεια και κατανόηση τις πιέσεις τις οποίες ε, αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και άλλα κράτη στον κόσμο που ε, αισθάνονται την ανάγκη και πιέζονται να αναλάβουν άμεση δράση και στην διάμεση ενδιάμεση έκθεση. Αυτό αναγράφεται. Βεβαίως ε, τα κράτη επιτρέπονται, επιτρέπεται στα πλαίσια του εσωτερικού δικαίου να ε, νομοθετούν όπω το επιθυμούν, αρκεί να είναι εντάξει με τι διεθνεί του υποχρεώσεις. Η μόνη βασική γραμμή στον ΩΣΑ είναι πως οποιαδήποτε μονομερής δράση αναλαμβάνει μια χώρα θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί με έναν τρόπο που δεν θα υποσκάφτει την πρόοδο την οποία εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε τη στιγμή που σχεδιάζουμε μια μακροπρόθεσμη λύση. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ λοιπόν έχουμε τις, ε, ε, την ευκαιρία να μιλήσουν και οι συνεισηγητές από την ΕΚΟΝ. Νταρίους, ναι. μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρχήν. Τα προβλήματα που ενδεχομένω θα δημιουργήσει η διάκριση μεταξύ ψηφιακών υπηρεσιών που θα φορολογούνται και άλλων ψηφιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν κάποια κράτη. Είναι εύκολο να γίνει αυτό σε κάθε περίπτωση και με σαφήνεια να ε, οριοθετηθεί δηλαδή έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαιές ζώνες όπου κανείς δεν θα γνωρίζει ποια είναι η φορολογητέα η υπηρεσία και ποια όχι για μένα δεν είναι τόσο σαφές, γιατί οι ορισμοί ακόμα είναι γενικόλογοι. Και σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως οι εθνικές φορολογικές αρχές είναι έτοιμες να κάνουν αυτή τη διάκριση και να μετρήσουν αυτές τις φορολογητές ψηφιακές υπηρεσίες. Είστε πεπισμένους πως έχουν τη δυνατότητα να το αξιολογήσουν αυτό και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις προτάσεις Επίσης έχω μία ερώτηση και στρέφομαι προς τον Όσα. Είναι λίγο συνέχεια της προηγούμενης ε, ερώτησης. Κάποια κράτη στον Όσα είναι κατά αυτής της φορολογίας, ε, τουλάχιστον είναι κατά της γενικότερης ε, έννοιας του ψηφιακού φόρου. Γιατί λοιπόν είναι εναντίον, ποια είναι τα επιχειρηματά τους και εσείς είστε ακόμα πεπισμένους πως θα βρείτε μία λύση συμβιβαστική μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια για να έχουμε μια μαγκόσμια λύση. Εάν ναι, τι είδου επιχειρήματα η τακτική προτείνεται για να πείσετε αυτού οι οποίοι δεν θέλουν να σας ακούσουν. Και δεν θέλουν καθόλου να σκεφτούν αυτή την ε, δυνατότητα. Επίσης, σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η μονομερής δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εγώ στηρίζω, βοηθά προς την εξέβρεση μιας παγκόσμιας λύσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει αυτή τη δράση με τούτο το εργαλείο μόνη της. Πιστεύετε πως αυτό παρακινεί τα άλλα κράτη προς μια κοινή λύση. Ή τα προκαλεί να αντισταθούν. Τι πιστεύετε. Είστε υπέρ των όσων κάνουμε εδώ αυτό τον οποίο ξεκινήσαμε μέσω της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω των δικών μας εκθέσεων. Ευχαριστώ πολύ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yeah, thank you for your question. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Η διάκριση μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, όπως τις περιγράφουμε και στην οδηγία, καταρχήν Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ στοχευμένη οδηγία που καλύπτει μόνο τρεις συγκεκριμένες δραστηριότητες και ουσιαστικά στην πράξη δεν έχει επιπτώσεις αυτό όσον αφορά την εφαρμογή του νομοθετικού αυτού κειμένου. Και βεβαίως ε, όσο λιγότερες ε, υπηρεσίες συμπεριλαμβάνει ένα κείμενο, τόσο πιο εύκολη είναι η εφαρμογή του. Και όσο περισσότερες, τόσο πιο πολλά προβλήματα προκύπτουν ως προς την εφαρμογή. Βεβαίως καταλαβαίνω αυτό που λέτε, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, όχι μόνο από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και από μέρους μεμονωμένων κρατών. Μπορούμε να διευκρινίσουμε και οι ερωτήσεις μας βοηθούν, ποιες φορολογικές υπηρεσίες ε, θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Είμαστε ανοιχτοί και δεχόμαστε σχόλια από μέρους σας εάν αυτά οδηγούν σε περισσότερη αποσαφήνιση και διευκρίνηση του κειμένου. Όσον αφορά τους ορισμούς, όπως σε κάθε νομικό κείμενο, ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολύ συγκεκριμένες έννοιες όπως οι εξαιρέσει. Τι παραδείγματο χάρη εξαιρείται, σε ποιες υπηρεσίες επιβάλλεται ΦΠΑ ή άλλη φορολόγηση για να μην γίνονται ε, λάθη και διακρίσεις. Και βεβαίως ε, έχουμε κάθε εμπιστοσύνη στις ε, φορολογικές αρχές των κρατών μελών, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος, ε, η εκτίμηση και να συμμορφωθούν με τα κείμενα όταν θα ψηφιστούν. Όσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά το πρώτο σημείο που αφορά το DST, γιατί κάποιες χώρες παραδείγματος χάρη συνεχίζουν να εκφράζουν ανησυχίες όσον αφορά την υιοθέτηση. Ένας από τους λόγους θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχουν ε, οικονομικές τρευλώσεις που ουσιαστικά απορρέουν από τέτοια μέτρα η κάθε μονομερής δράση, η κάθε εθνική δραστηριότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται, να συνάδει με τις διεθνείς αρχές που φυσικά συμπεριλαμβάνουν την αρχή της μη διάκρισης και φυσικά και όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό είναι αν θέλετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει περιθώριο ελιγμού. Η κάθε χώρα μπορεί να σχεδιάσει τα δικά της μέτρα τα οποία να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στη δικέ στις δικές της ιδιαιτερότητες, ε, στα χαρακτηριστικά της δικής της οικονομία. Κάτι άλλο που ακούσαμε από άλλες χώρες είναι ότι οι μακροπρόθεσμες λύσεις θα πρέπει να βρεθούν με προθεσμία το 2020 και το ερώτημα αν ε, αξίζει να υιοθετηθούν σήμερα προσωρινά μέτρα, γιατί το 2020 είναι πραγματικά και βάση των ε, διαδικασιών του ΟΣΑ, αλλά και οι νομοθετικές διαδικασίες των κρατών μελών είναι τόσο χρονοβόρες που το 2020 είναι αύριο το πρωί. Είναι πάρα πολύ μικρή ε, στενή προθεσμία. Υπάρχει λοιπόν λόγος προσωρινών μέτρων, αλλά όσον αφορά μονομερή άμεση δράση τύπου DST ή άλλα μέτρα σε αντιπαράθεση με μακροπρόθεσμες λύσεις και μέτρα, σίγουρα κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτών των μακροπρόθεσμων μέτρων τα έχουμε ήδη συζητήσει, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρξει μια ρήτρα προθεσμίας ή ε, ημερομηνία λήξης όσον αφορά δηλαδή την λήξη αυτών των μέτρων σε περίπτωση που τελικά υιοθετηθούν, συμφωνηθούν ε, μακροπρόθεσμες λύσεις σε διεθνές επίπεδο. Κάποιες χώρες μπορεί να θεωρήσουν ότι η πρόταση για υιοθέτηση μονομερών ε, μέτρων μπορεί να είναι κάτι χρήσιμο, έτσι ώστε να πιεστούν άλλες χώρες για να υπάρξει συμβιβασμός και για να υπάρξει σύγκληση, μέτρα σύγκλησης και βήματα προς την κοινή κατεύθυνση. Αυτό για μένα είναι κάτι το πολιτικό, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ευχαριστώ. Έχουμε 8 ομιλητές που αντιπροσωπεύουν πολιτικές ομάδες. Πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των ερωτήσεων και να βραχύνουμε στο τετράλεπτο το χρόνο παρέμβασης. Εκτός μικροφώνου συζήτησης. some... Και για κάποιους άλλους υπήρχε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που διατέθη, αλλά ήταν συνεισηγητές. Ήταν κάτι διαφορετικό. Τέλο πάντων. Ότμαρ Κάρας για το ΕΛΚ. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Δεν μιλάμε μόνο για θέματα που αφορούν, ε, αν θέλετε, επιχειρήσεις, ε, με ύποπτες πρακτικές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο σημαίνει και εντός υπάρχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ξέρετε πολύ καλά ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο ΕΚΟΦΗΝ συζητήθηκαν τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα θα πρέπει να ξαναδεί τον κανόνα της ομοφωνίας για τέτοιου είδους θέματα, κάτι που πραγματικά εμποδίζει αποτελεσματικές αποφάσεις. Επίσης το θέμα της α, κακής θα έλεγα οριοθέτησης του ψηφιακού και μη ψηφιακού κόσμου στην οικονομία. Θα πρέπει να δούμε λίγο και τα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα. Για μένα το ιδανικό θα ήταν αυτά να είμαι σε ένα μείγμα, γιατί εδώ μιλάμε για το 3%, μιλάμε για δισεκατομμύρια, για το 3% της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα έσοδα, οι ίδιοι πόροι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Yes, the commission, please, Mr. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Φόσακας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σας, κάναμε μια πρόταση αναφέρεστε στον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών και τα προσωρινά μέτρα. Κάναμε πρόταση βάσει του άρθρου 113 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί ομοφωνία. Αυτό είναι το ενδεχόμενο που επεξεργαζόμαστε. Για τη δεύτερη ερώτηση. Ψηφιακές υπηρεσίες, μη ψηφιακές, διάκριση τίθεται στο θέμα της συζητήσεως. Τι αποτελεί ψηφιακή υπηρεσία, τι όχι. Είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να μείνουμε εκτός αυτής της συζητήσεως. Πώς. Καθορίζοντας κάποιες υπηρεσίες συγκεκριμένες και τα χαρακτηριστικά αυτών. Αυξήσαμε την ασφάλεια δικαίου ο τρόπο για τι εφοριακέ αρχέ και τι επιχειρήσει όσον αφορά την ταξινόμηση δραστηριοτήτων στον πραγματικό κόσμο. Και ποιε δραστηριότητε είναι αυτέ που πρέπει να φορολογηθούν από τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Ζητώ συγγνώμη αν δεν απαντώ έτσι στην ερώτησή σα. Πείτε το μου. Μετά, η δυνατότητα που υπάρχει να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από τον ψηφιακό, το φόρο ψηφιακών υπηρεσιών για τους ιδίους πόρους. Στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνοδεύει το ψηφιακό φόρο και το σχετικό πακέτο γινόταν μενία αυτής της δυνατότητας. Από ό,τι γνωρίζω, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί εκτενώς το συγκεκριμένο θέμα που θέσατε. Schlein. Κυρία Σλάιν, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάλεξε το 3% για αυτό το προσωρινό ψηφιακό φόρο. Μετά από σεχτική ανάλυση διαφόρων παραγόντων, λέει, και αντιχτύπου, βάρους φορολόγησης των επιχειρήσεων με διαφορετικά περιθώρια κέρδους. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε περισσότερο αυτό που προανέφερα, που είπατε. Άλλη ερώτηση. Πόσες εταιρείες όλο τον κόσμο είδε τα στοιχεία που αναφέρετε στην παρουσίασή σας. Έχετε κάποια ιδέα πόσες εταιρείε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως φορολογήσιμα πρόσωπα σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 4. Τελευταία ερώτηση. Αυτό πώς ταιριάζει με την απαιτούμενη διαθροτική απάντηση κοινοδηγία CCTB. Μήπως έτσι καθυστερεί η, έγκριση του CCTB. Και από αυτού το Κοινοβούλιο επανειλημμένα μεγάλη πλειοψηφία θεώρησε και εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη Καταρχάς, διότι η ομάδα που εξεργάστηκε το θέμα είναι αρκετά πολυμελής. Δεν μείνατε δυστυχώς με τους οικονομολόγους της ομάδας και συγχωρήστε μας για τις βασικές εξηγήσεις που θα σας δώσουμε. Με τα χαράς να διαβιβάσουμε ε, τυχόν γραπτές ερωτήσεις αργότερα και στο βαθμό του δυνατού να διευκρινίσουμε τις απορίες. Το 3% αυτό αποφασίστηκε ούτως ώστε να εξισορροπηθεί η ανάγκη συλλογής εισοδημάτων για να αντισταθμιστούν οι δαπάνες στην εφαρμογή του μέτρου και απ' την άλλη παραδεχόμενοι το ότι αυτός ο συμπληρωματικός φόρος πιθανότατα θα δημιουργούσε στρεβλώσεις στην περίπτωση κατά την οποία οι εταιρείε που πληρώνουν τον ψηφιακό φόρο ε, ταυτόχρονα υπόκεινται και σε φόρο ε, εταιρικό σε ένα κάτω Διάφορα περιθώρια λήφθησαν υπόψη και οι, οι, που θα υποστούν τη διπλή φορολόγηση αυτή είναι κάτι που έχει υπολογιστεί. Ποσοστό πάνω από 3% οδηγούσε σε επίπεδα φορολόγησης που θεωρήθηκαν ότι παρεμποδίζουν και παρενοχλούν σε σημαντικό βαθμό τη βιωσιμότητα των εταιριών αυτών. Ενώ χαμηλότερος φόρος, χαμηλότερο ποσοστό φορολόγησης δεν εξασφάλιζε την οικονομική βιωσιμότητα του φόρου αυτού καθεαυτού. Γι' αυτό 3% κατά την άποψη της ήταν ένα συμβιβασμό μεταξύ των δύο προαναφερθησών πτυχών που χρειαζόταν εξισορρόπηση. Για δεύτερη ερώτηση, εκτιμούμε ότι περίπου 180 με 200 εταιρείε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να υποστούν αυτό το φόρο του ψηφιακών υπηρεσιών. Είναι εταιρείε που ξεπερνούν τα δύο όρια και που παρέχουν φορολογητέ υπηρεσίε. Και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Όσον αφορά το CCTB, βάσει τη προτάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το CCTB δεν εφαρμόζεται όλε τι εταιρείε, διότι υπάρχει πρέπει να έχουν τουλάχιστον 750 εκατομμύρια ευρώ εισόδημα για να, μπουν σε αυτό το πλαίσιο εταιρείε. Αν εγκριθεί το CCCTB και πάλι χαζόμαστε κανόνες για άλλε εταιρείε που δεν υπόκειται στους κανόνες του CCCTB. Τούτου λεχθέντο. αναγνωρίζουμε πράγματι ότι οι προτάσεις για την κοινή βάση και το CCCTB θα πρέπει να προσαρμοστούν εν ευθέτω χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την ψηφιακή παρουσία και θα πρέπει να προσαρμόσουμε δεόντως τους τύπους περικατανομής. Και το Ευρωκοινοβούλιο έκανε ενδιαφέρουσε ε, προτάσει σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σλάιν γιατί κάνατε πολύ καλή ερώτηση σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ε, από του φιλελεύθερου ο συνάδελφο, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη τύχη και δεν καταφέραμε εύκολα να βρούμε βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει ε, σε θέματα φορολογικά. Γιατί λοιπόν πιστεύετε πως ε, αυτή τη στιγμή ο φόρος της υπηρεσίας, ψηφιακής υπηρεσίας θα έχει καλύτερη τύχη τι θα γίνει, θα έχουμε την ίδια τύχη με τον φορό για τις ε, συναλλαγές, νομίζω θα χρειαστεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και θα φορολογούμε τα κέρδη ή τον κύκλο εργασιών έτσι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε και κάποια κέρδη τα οποία δεν εμφανίζονται ε, δεν φοβόσαστε εσείς ε, τι θα γίνει και αν θα πάρουν αντίματρα αυτές οι εταιρείε, οι κολοσσοί, οι αμερικάνικες, οι οποίες είναι οι βασικές που θα φορολογηθούν. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί ο φόρος αυτός της ψηφιακής υπηρεσίας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά με πολύ πιεστικές προθεσμίες για να σχεδιάσουμε τρεις προτάσεις και μία πλήρη επιδοσιολογική μελέτη, οι οποίες να είναι σε τεχνικά ε, στέρεη βάση και αναγνωρίζουμε πως μας έχει ασκηθεί κάποια κριτική, ξέρουμε ποια είναι αυτή, αλλά θέλω να τονίσω πως δεν έχω ακούσει να υπάρχουν σοβαρές εναλλακτικέ λύσεις προτάσεις που εμείς έχουμε καταθέσει. Αυτό πρέπει να το δούμε. Θέλουμε να είναι τεχνικά βάσιμες οι προτάσεις μας όταν τις καταθέσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να λαμβάνουμε υπόψη αφού ακούσουμε οποιασδήποτε λογικές προτάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να δώσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερη ποιότητα σε αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Γιατί δεν κάνουμε φορολόγηση σε κέρδη και σε εισόδημα και κάνουμε ε, προσπάθεια φορολόγηση κύκλου εργασίας. Ε, δεν είναι αυτό που επιθυμούμε, αλλά ελείψη μιας ε, παγκόσμιας λύσης, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, θεωρούμε πως μια ευρωπαϊκή αλλαγή των κανόνων για την εταιρική φορολογία, δηλαδή κάτι που συνδυάζει τα έσοδα και το κέρδος και φορολογία αυτά από κοινού θα είναι η καλύτερη δυνατόν επιλογή. Όμως θα πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικές, ουσιαστικές ε, πτυχές του, ε, της φορολογίας επιχειρήσεων. Οπότε εντωμεταξύ χρειαζόμαστε κάποια διάμεσα μέτρα ε, τα οποία θα ασκήσουν όσο συζητάμε, θα, θα εφαρμόσουμε όσο συζητάμε τις παγκόσμιες λύσεις. Είπαμε, παγκόσμιος φόρος στις, ε, στον όγκο συναλλαγών και όχι στα κέρδη, γιατί διαφορετικά αν μείνουμε στη φορολόγηση των κερδών θα παραμείνουμε στο ίδιο επιχειρηματικό πλαίσιο, φορολογικά επιχειρηματικό πλαίσιο, στο οποίο προσπαθούμε να αλλάξουμε, δίνοντας μια μακροπρόθεσμη λύση. Οπότε ως ενδιάμεσο μέτρο προτείνουμε κάτι διαφορετικό και όχι κάτι το οποίο τρίτον στις κατηγορίες της κλασικής φορολογίας ε, επιχειρήσεων. Για την τελευταία ερώτηση για αντίπινα και αντίπινα δεν μπορώ να πω ότι θα κάνω άλλες δικαιοδοξίες. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω για φορολογία ε, πάνω σε επιχειρήσεις, σε ομάδες επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεων από συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Είναι σφαίρνει αυτές τις ψηφιακέ υπηρεσίες από όπου και να προέρχεται και όπου και να είναι εγκατεστημένη. Thank you. The Greens have Πολύ. Ευαζολή για τους πράσινους. Θα ήθελα να κάνω ερώτηση στον εκπρόσωπο του ΩΣΑ εάν προσπαθείτε να διορθώσετε κάτι το οποίο δεν ε, διορθώνεται την ε, πρόσφατη παρουσίαση που κάνετε ότι παρόλο τους καινούριους κανόνες παρόλη τη νέα διακυβέρνηση, παρόλες τους νέους κανόνες το αποτέλεσμα είναι αποτυχία. Δαπανίσατε χρήματα, χρόνο, σειρά, προσπάθειες το είναι ότι υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν τεράστια κενά στη φορολόγια, ακόμα και χώρες όπως η Βραζιλία. κανόνες βλέπουμε και άλλες χώρες